I think we will make a start. Um, apologies for being late, but as you all know there is... Καλημέρα συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, όμως όπως γνωρίζετε σήμερα στις Βρυξέλλες ε, υπάρχει μια απεργία και η εισηγήτρια δεν έχει μπορέσει να έρθει ακόμα, ωστόσο πρέπει να ξεκινήσουμε την ακρόαση γιατί είναι πολύ σημαντική. να συζητήσουμε, όπως γνωρίζετε, για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία. Ένα θέμα κρίσιμο, κρίσιμη σημασία. Γιατί δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα οι γυναίκες που, έχουν και αναπηρία, που είναι επίση άτομα με αναπηρία. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Πρόσφυγες, μπορεί να ε, μιλούμε για πολλές διαφορετικές μορφές αναπηρίας και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές μορφές διακρίσεων επίσης σε θεσμικό επίπεδο, σε πρακτικό επίπεδο, στην αγορά εργασίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα. Ο Οργανισμός των Εθνών με το, την συμφωνία, συγγνώμη, το Σύμφωνο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται αυτές οι γυναίκες και καλεί από τα κράτη που έχουν υπογράψει αυτό το σύμφωνο να ε, αναλάβουν δράση, να εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών ε, των ατόμων αυτών. Πιστεύω και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε ότι με την ακρόαση μας σήμερα θα βοηθηθούμε στην προετοιμασία της ε, έκθεσης που ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και προετοιμάζει η συγγήτρια της Επιτροπής μας, η οποία όπως σας είπα δυστυχώς δεν προφτάσει να έρθει στη συνεδρίαση. Γι' αυτό προτείνω να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές και όταν έρθει η συγγήτρια θα της δώσω το λόγο. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο ομιλητή, την πρώτη ομιλητρία από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, η κυρία Πελάης. The mic, please. Okay, thank you. Thank you so much. I will speak in Spanish. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα ισπανικά αν δεν σας πειράζει. Φορέστε λοιπόν τα ακουστικά σας, λέει ο μιλήτρια. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα σας, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Ονομάζομαι Άννα Πελάιθ Ναρβάιθ και εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ανθρώπων με Αναπηρία που είναι η ευρωπαϊκή ομπρέλα δομή όλων των οργανισμών και ενώσεων που εκπροσωπούν ε, στην ε, περιφέρειά μας ανθρώπους με αναπηρία. Αυτή τη στιγμή 85 εκατομμύρια πολίτες έχουμε, εκ των οποίων το 60% περί τα 51 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία. Προσωπώ επίσης ε, το Ίδρυμα Θέρμη Γυναίκες που έχει μια επιτροπή εκπροσώπησης των γυναικών με αναπηρία προκειμένου να μεταφραστεί στην πρακτική η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία στη χώρα μου, την Ισπανία. Έχουμε 2017, λέει ο Μιλήτρια και επομένως εορτάζουμε 20 χρόνια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ υπάρξεως και πολλά από τα εθνικά συμβούλια όπως το δικό μας το Θέρμη για εκπροσώπηση δηλαδή ανθρώπους με αναπηρία που φέτος μάλιστα το Θέρμη θα λάβει και το Ευρωπαϊκό Βραβείο σε αυτά τα χρόνια που έχουν παρέλθει πολλά έχουν γίνει έχουμε πετύχει κάποιες βελτιώσεις, έχουμε μια συνθήκη επικυρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των 51 αυτών εκατομμυρίων πολιτών. Έχουμε ένα θεματολόγιο ανάπτυξης 2030 με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τους ανθρώπους με αναπηρία στα θέματα τόσο σημαντικά όσο είναι η παιδεία και η εργασία. Έχουμε προχωρήσει αλλά μας μένουν πάρα πολλά ακόμα να κάνουμε. Όμως ποια είναι η θέση των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία που έχουν μείνει στο μεσοδιάστημα πως έχουμε εξασφαλίσει τα θεμελιώδη τους δικαιώματα διότι είναι βέβαιο πρόεδρε συνάδελφοι, ότι οι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία εξακολουθούν σήμερα να υποφέρουν. Σήμερα, εν έτη 2017, από έντονη φτώχεια, από διάφορες παραβιάσεις εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και πολύ συχνά η μόνη μορφή, η μόνη λύση επιβίωσης είναι είσοδο σε διάφορα ιδρύματα. Υπάρχει συνεχιζόμενος αποκλεισμός από την αγορά εργασίας από τους αντίστοιχους άνδρες με αναπηρία ή τις υπόλοιπες γυναίκες. Οι γυναίκες με αναπηρία αποκλείονται από την κοινωνία της πληροφορίας, αποκλείονται από τις υπηρεσίες που αφορούν γενικά στις γυναίκες συμπεριλαμβανομένων κάποιων συγκεκριμένων ειδικών υπηρεσιών για ανθρώπους με αναπηρία. Δυστυχώς, δεν μπορούν να ασκήσουν και τα γενετικά τους ακόμα δικαιώματα, διότι έχουν αναπηρία. Δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε πολλές περιπτώσεις έχουν ε, περιορισμό στη δυνατότητα τους νομικής εκπροσώπησης. και πολύ σημαντικά ποσοστά των γυναικών αυτών δεν θα μπορούν να ψηφίσουν. Δεν μπορούν και δεν θα μπορούν, διότι δεν έχουν τη νομική δυνατότητα κατόπιν διαδικασιών αμβλώσεων αναγκαστικών ή άλλων γενετικών επιθετικών παρεμβάσεων έχουν απολέσει τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν τις προσωπικές τους αποφάσεις, τις αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους τον εαυτό τους. Έχουμε λοιπόν μια σειρά, σειρά από διαρκείς προκλήσεις και προβλήματα, ώστε αυτές οι γυναίκες να μπορούν να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους. Και πρέπει να έχουμε μια διπλή αστίαση απέναντι στο πρόβλημα αυτό. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, τις πολλαπλές διατομιακές διακρίσεις που υφίστανται εδώ και δεκαετίες και αιώνες αφενός και αφετέρου πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις βοηθήσουμε να ενταχθούν πιο πλήρως στην κοινωνία και στην αγορά το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε νομοθεσίες και πρακτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Ώστε να μην έχουμε διακρίσεις επί τη βάση του φύλου. Ή ώστε να καταγράφονται τα σεξουαλικά εγκλήματα που υφίστανται πολλές από τις γυναίκες αυτές με συγκεκριμένο νομικό τρόπο. Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές αυτέ διακρίσει, πρέπει να υιοθετήσουμε διατάξεις και μέτρα επαρκή ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαφοροποίηση δικαιωμάτων που υφίσταται. Να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια που αποτρέπουν τις γυναίκες με αναπηρία από το να έχουν την εγγύηση ότι η φωνή τους θα ακούγεται σε θέματα που τις αφορούν άμεσα όπως και στην παρακολούθηση και τον σχεδιασμό των πολιτικών. Χρειάζεται να αναλύσουμε και να αναλύουμε δεδομένα επί της προσωπικής κατάστασης πολλών γυναικών σε διάφορα πεδία που αφορούν στη ζωή των γυναικών με αναπηρία. Οποιαδήποτε πολιτική αφορά γενικώ τις γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις αναπηρίες. Αντιστοίχως προς οποιαδήποτε πολιτική συγκεκριμένη για τις αναπηρίες, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη της συγκεκριμένα τον πληθυσμό των γυναικών με αναπηρία. Η ισότητα των φίλων αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνει υπόψη της την ιδιαιτερότητα των αναγκών των γυναικών με αναπηρία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να εξασφαλίσουμε τη συμπερίληψη του πληθυσμού αυτού ενεργώς στις πολιτικές ε, συνεργασίας και ανάπτυξης στο θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καταρχάς θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμείνουμε εδώ ώστε να καταργήσουμε τις διατάξεις αυτές που αποτρέπουν την ίση συμμετοχή των γυναικών αυτών στην ε, δημόσια ζωή, στο δημόσιο βίο έχουμε συγκεκριμένο πληθυσμό στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες 51 εκατομμύρια συνολικά όχι στο συγγνώμη λέει η ομιλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 60% έχουμε από τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα ψήφου είναι γυναίκες με αναπηρία λέει περίπου η ομιλήτρια πρέπει να συνεχίσουμε εν πάση περιπτώσει να βοηθούμε τις γυναίκες και τα κορίτσια αυτά με συγκεκριμένα μέτρα για να εξασφαλίζουμε την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη, στην εργασία ώστε να μην έχουμε κρούσματα βίας. Έχουμε την ε, σύμβαση της Ισταμπούλ που έχει επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει στην πράξη να προχωρήσουμε σε μέτρα και διατάξεις την υγεία, την οικογενειακή, την ε, γενετική, την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένα δίκτυα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία. Πριν από 20 χρόνια με το Έλιος 2 έργο ξεκινήσαμε για τους ανθρώπους με αναπηρία 20 χρόνια αργότερα θα πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, όπου μόλις 7 χώρες έχουν συγκεκριμένο φορέα, οργανισμό που εκπροσωπεί τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία. Χρειάζεται επίσης υποστήριξη για την υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων ώστε να εξασφαλίζονται τα νομικά και πολιτιακά τους δικαιώματα, ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία να μπορούν να λάβουν τις προσωπικές αποφάσεις που αφορούν στη ζωή τους. Πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να υπερβούμε τα εμπόδια που υφίστανται για τις διακρίσεις αυτές με την άμεση συμμετοχή του πληθυσμού των γυναικών και κοριτσιών που έχουν το πρόβλημα. Χρειάζεται συστηματική επίσης υποστήριξη σε τεχνική αρρωγή μέσω διεθνούς συνεργασίας και σε άλλες χώρες ώστε να βοηθήσουν τους αντίστοιχους δικούς τους πληθυσμούς. Και σκεπτόμενοι τις γυναίκες με αναπηρία θα σκεφτόμασταν ένα πληθυσμό αντίστοιχο των χωρών της Σουηδίας, του, της Ολλανδίας, του Βελγίου ή της ε, Ελλάδος δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεχνούμε ολόκληρους τέτοιους πληθυσμούς που ισοδυναμούν με τις χώρες που σας ανέφερα. Αλλά το κάνει για τον πληθυσμό των συνολικών των γυναικών με αναπηρία. Ποιους λοιπόν έχουμε αφήσει πίσω. Η απάντηση είναι σαφής. Τις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα εξερτάται να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλος, με, μέλλον με για τις γυναίκες αυτές. ευχαριστούμε πολύ την Άννα. Ιδιαίτερα σημαντικά σημεία έθιξε στην ομιλία σου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση ήταν τόσο θλιβερή σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ψήφου των γυναικών με αναπηρία. Βεβαίω είναι κάτι που θα πρέπει να μα ανησυχεί, καθώ και όλα τα υπόλοιπα σημεία που έθιξε. Πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φούλων που θα μας μιλήσει για την αποδοχή και θα μας εξηγήσει λίγο καλύτερα τι ακριβώς κάνει. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ διάφορους συνδέσμους που υποστηρίζουν γυναίκες και παιδιά με προβλήματα νοηματικής αναπηρίας. και θέλουν να μπορούν να εκφράζουν μια άποψη τέτοια για την κατάστασή τους τα άτομα αυτά. Βεβαίως η κατηγορία αυτή άφορα και γυναίκες και παιδιά που έχουν προβλήματα διανόησης και πάντα βρίσκονται στα, περιθρό, στα περιθώρια τόσο τα μικρά παιδιά, τα μικρά κορίτσια, όσο και οι μητέρες τους που σε πολλές περιπτώσεις είναι υποχρεωμένες να στηρίζουν τα παιδιά με αυτά τα προβλήματα. Η Άννα έθιξε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα άτομα με αναπηρία. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να κάνω κάποιες συγκρίσεις. Τα άτομα που έχουν διανοητικά προβλήματα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει κάποιοι άλλοι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αντικείμενα βίας, φυσικής βίας, ε, εκμετάλλευσης. Οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν προβλήματα διανοητικής αναπηρίας δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό, είναι, να τον εαυτό τους, είναι ακόμη πιο ευάλωτα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες και τα παιδιά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και προσπαθούν να εργαστούν ώστε να απολαμβάνουν ε, και αυτά τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι όπως αναγνωρίζονται, παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. ούτω ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την αυτονομία των γυναικών έχουν α, ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε το στόχο αυτό, υπάρχουν κάποιες δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Η συνειδητοποίηση αυτή βεβαίως πρέπει να γίνει σε επίπεδο ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Έχουμε στην... Στις Βρυξέλλες είχαμε το, το Σαββατοκύριακο του Μαραθώνα, του ε, Μαραθώνιου, με συγχωρείτε, την προηγούμενη εβδομάδα. Ο νικητής κέρδισε ένα εκατομμύριο. Χίλια ευρώ. Με συγχωρείτε. Ε, η γυναίκα, ε, η γυναίκα νικήτρια κέρδισε πολύ λιγότερα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό. Είναι ανάγκη να υπάρξει μια εκπαίδευση που θα επιτρέψει στα άτομα αυτά να πάρουν τον έλεγχο της δικής τους ζωής. Θα τους επιτρέψει επίσης να αντισταθούν στις διακρίσεις και στην εκμετάλλευση. Πρέπει επίσης, όπως είπε και η Άννα, να υπάρξει μια νομική προστασία αποτελεσματική των γυναικών και των κοριτσιών που δεν μπορούν να εξασκήσουν ούτε καν το νομικό τους δικαίωμα της ψηφοφορίας. Πρέπει να υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές και νόμοθεσίες που θα εγγυώνται σε οποιαδήποτε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων τους ή εκμετάλλευσης θα μπορούν να αντιδράσουν νομικά. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σεβασμό σε ό,τι αφορά τις αναπαραγωγικές, τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Σήμερα τα άτομα με διανοητική υστέρηση, γυναίκες με διανοητική υστέρηση και τα μικρά κορίτσια δεν έχουν πρόσβαση σε μια φυσιολογική αναπαραγωγική ζωή. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα και αυτά τα άτομα να σχεδιάζουν ε, την οικογενειακή του ζωή. Στο Βέλγιο υπήρχε ένας νόμος που προστάτευε τα άτομα με διανοητική αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία γενικά. το οποίο δημιουργού, ένας νόμος που δημιουργούσε διάφορα προβλήματα στα άτομα αυτά. σε ό,τι αφορά τα ίσα δικαιώματα που έχει ένα άτομο χωρίς αναπηρίες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία, είναι ανάγκη να ευαισθητοποιηθούμε όλοι απέναντι σε αυτά τα άτομα με διανοητική στέρηση, στις γυναίκες και στα μικρά κορίτσια. Και τι συμβαίνει λοιπόν σε ό,τι αφορά τις μητέρες είναι μητέρε που δεν καταφέρνουν να έχουν μια επαγγελματική ζωή, μια φυσιολογική οικογενειακή ζωή γιατί είναι υποχρεωμένε να στηρίζουν αυτό το παιδί με διανοητική υστέρηση το οποίο ακόμη και όταν θα γίνει ενήλικας μπορεί να μην έχει απαραίτητα την στήριξη που του χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να αποφύγουμε τις διακρίσεις κατά βάρος αυτών των γυναικών που γίνονται και αναγκαστικά καθώς είναι υποχρεωμένες να στηρίζουν τα παιδιά τους τις διακρίσεις που συμβαίνουν κατά συνέπεια. Να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών αυτών που έχουν πάψει να εργάζονται, που πολλές φορές δεν έχουν καν ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας να τις προστατεύει και είναι υποχρεωμένες να στηρίζουν τα παιδιά τους χωρίς να έχουν καμία απολύτως οικονομική αποζημίωση. Αυτό που πρέπει να σας πω, το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι όλοι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και αυτό το δρόμο προσπαθούμε να διανύσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ λέει η Πρόεδρος. Εξαιρετικά διαφωτιστική η ομιλία σας. Πράγματα που δεν είχαμε λάβει υπόψη μας προηγουμένως ίσως. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βαν από τον Οργανισμό Εκπαίδευσης Χωρίς Αποκλεισμούς και θα μιλήσει Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και την Επιτροπή για την πρόσκληση. Είμαι συντονίστρια του φορέα υποστήριξης των γυναικών με, με, με, των ατόμων με αναπηρία και θα ήθελα να προσθέσω ορισμένου προβληματισμού, εστιάζοντα κυρίω στο ζήτημα τη εκπαίδευση και τη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Έχω προετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint, αν μπορούμε να την ε, δούμε, για να παρακολουθείτε καλύτερα την παρουσίασή μου. Φυσικά δεν θα σταθώ μόνο στις διαφάνειες. Θα σας μιλήσω για τις δραστηριότητες του οργανισμού μας, παρέχει γενικότερε υπηρεσίε υποστήριξη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη Βαλονία και στη Φλάνδρα. Προσπαθούμε δηλαδή να βοηθήσουμε ε, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση των ε, ατόμων με αναπηρία στα, στα πανεπιστήμια. Έρχεται σιγά σιγά εκεί. Παρουσίασή μου, ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, όπως σας είπα, οι προσπάθειες δικές μας εστιάζονται στο να ε, υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη πρόσβαση ε, των φοιτητών με αναπηρία. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε με θεσμικές παρεμβάσεις, να, με επικοινωνία με τους αρμοδίους στα πανεπιστήμια έτσι ώστε να καταπολεμηθεί ο αποκλεισμός και να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν αυτή την πρόσβαση. ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία, που είναι και το θέμα συζήτησης σήμερα. Το 16% των γυναικών στην Ευρώπη είναι γυναίκες με αναπηρία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία της ισότητας των δύο φύλων. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα τους και τις γυναίκες με, ε, αναπηρία, ε, με αναπηρία. Όμως αυτός είναι ο πληθυσμός και φυσικά υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Το άρθρο 6 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία αναφέρεται συγκεκριμένα σε δικαιώματα, για, συγγνώμη, σε μέτρα για την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η κοινωνική ομάδα πλήττεται εξαιτίας πολλαπλών διακρίσεων. και Αντίστοιχε προβλέψει υπάρχουν και στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ευτυχώ τα κράτη-μέλη έχουν προσπαθήσει να πάνε, ένα, να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Και υπάρχουν λοιπόν εθνικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την βελτίωση τη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασία και στην εκπαίδευση, χωρί όμω δυστυχώ ακόμα να υπάρχει μια ε, συνολική ευρωπαϊκή οδηγία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην οποία βασιζόμαστε είναι η οδηγία 2078 για τον τομέα της εργασίας. Ωστόσο, ε, κοιτώντας τις διάφορες αναφορές, τη βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών με αναπηρία συνεχίζονται. και θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τι θα πρέπει να γίνει κατά τομέα. Ας ξεκινήσουμε από την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εδώ μας ανησυχεί η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στο χώρο εργασίας, γιατί δεν βρίσκουν ε, δουλειά, ε, υφίστανται διακρίσεις στην αναζήτηση εργασίας και εξαιτία του φίλου τους και εξαιτία της αναπηρίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ε, μικρότερη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Όπως σας είπα λοιπόν, έχουν να αντιμετωπίσουν δύο ε, ειδών διακρίσεις και εξαιτία του φύλου και εξαιτία των ε, της αναπηρίας τους. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα των γυναικών να εργαστούν. Ε, υπάρχουν διαφορές στο ποσοστό ανεργία από χώρα σε χώρα, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση. Θα έρθουμε λοιπόν στο ζήτημα της εκπαίδευση. Και εδώ υφίστανται διακρίσει οι γυναίκε με αναπηρία αν και σε αυτόν τον τομέα οι διακρίσει σχετίζονται κυρίως με το, την αναπηρία και λιγότερο με το φύλλο, γιατί γενικότερα οι διακρίσεις εξαιτία του φύλλου στην εκπαίδευση είναι λιγότερο σημαντικές. Δεν έχουμε αρκετά στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μας για να γνωρίζουν ακριβώ ποια είναι η θέση των ε, γυναικών με αναπηρία στο, στο χώρο τη εκπαίδευση. Τα συστήματα παρακολούθηση που υπάρχουν πρέπει δηλαδή να βελτιωθούν. Θα σα δώσω ορισμένα στοιχεία που έχουμε εμεί στη διάθεσή μας. Ε, δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο σημαντική είναι η ε, ύπαρξη στατιστικών στοιχείων. Τα στοιχεία που σας δείχνω προέρχονται από ένα πανεπιστήμιο στη Φλάντρα. Η δικιά μας οργάνωση προσπαθεί να συλλέγει αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα για την κατάσταση των γυναικών με αναπηρία. Όμως, ακόμα δεν, τα έχουμε, δεν το έχουμε καταφέρει. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι η φοιτητέ με αναπηρία, αν του δούμε σε σχέση με το ποσοστό που, είναι τα, που έχουν τα άτομα με αναπηρία στο γενικό πληθυσμό, δεν ε, έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτό το πανεπιστήμιο επαρκώ. Αυτό είναι δικαιολόγητο. Γνωρίζουμε ότι ε, τα άτομα με αναπηρία ε, έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να, να επιτύχουν επιδόσεις ισότιμες με οποιονδήποτε άλλον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μερικές φορές ακόμα καλύτερες έχουν κάποια ιδιαίτερα ε, ικανότητε. και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να, τις, να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία να βρουν το, την κλίση τους και να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες τους. Βέβαια τα στοιχεία που σας δείχνω τώρα προερχόνται από ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο στη Φλάντρα, Όμως όπως σας είπα δεν έχουμε μια συνολική εικόνα. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε ποιες είναι οι βελτιστές πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν και άλλα πανεπιστήμια ή πού είναι τα προβλήματα και πού πρέπει να εστιάσουμε τις δράσεις αντιμετώπισης τους. έχουμε και άλλους τομείς πέρα από την εργασία και την παιδεία. Για παράδειγμα, η κατάσταση στο σπίτι, στην οικογένεια. Και εδώ έχουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία που δεν μπορούν πάντοτε ελεύθερα να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο προσωπικός τους ρόλος στα πλαίσια ας πούμε της ε, παιδείας που δίδεται στο σπίτι, στα πλαίσια επίσης της αντιμετώπισης κρούσματων βίας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αν σκεπτούμε από εκεί και πέρα και τον ελεύθερο χρόνο, την αναψυχία και εδώ έχουμε χαμηλότερη, πιο περιορισμένη συμμετοχή. Ποιε λοιπόν είναι οι συστάσεις που μπορούν να προκύπτουν. Είναι σημαντικό να θυμίζουμε ότι η αναπηρία έχει επιπτώσεις αντίκτυπο σε μια σειρά από παιδεία δραστηριότητας και για τους άνδρες και για τις γυναίκες βεβαίως, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτηρότητες της ε, διαφοράς των φύλων. Και είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας στους διάφορους τομείς τους παράγοντες αυτούς. Γιατί πολύ συχνά πρόκειται για μειονεκτήματα πολλαπλών επιπέδων στην πραγματικότητα. Και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να προχωρήσουμε σε μια σειρά ακόμα από μελέτες προκειμένου να έχουμε ασφάλεια δικαίου μεταξύ έλων ή μάλλον καλύτερη ασφάλεια δικαίου. Σας μίλησα για την οδηγία 78 του 2000 στο χώρο της εργασίας και στην περιοχή των αναπεριών. Πρέπει να εξετάσουμε και να προσέξουμε αυτούς τους πολλαπλούς ε, παράγοντες διακρίσεων. Και θα χρειαζόταν όλα αυτά να κωδικοποιηθούν σε μια οριζόντια οδηγία. Δηλαδή χρειάζεται προκειμένου να προετοιμάσουμε μια τέτοια νομοθετική πρόταση, ε, μια μελέτη που θα αποτυπώνει τις αναπηρίες σε όλες τις περιοχές σε όλα τα παιδεία και όχι μόνο στο εκπαιδευτικό. Επομένως ε, το δικό μας Ινστιτούτο εστιάζεται και στην σωστή απεικόνηση του προβλήματος, τη σωστή χαρτογράφηση του προβλήματος. Σε επίπεδο κοινωνίας πρέπει κανείς να έχει αντιληφθεί τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες αυτές. Η διελέχθη ότι έχουν γίνει μελέτες επί των φύλων και επί των αναπηριών, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάδραση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και τους σπουδαστέ με αναπηρίες. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, περισσότερα στοιχεία. Και για την ανώτατη εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό και εν ώψη της εισαγωγής τους στην αγορά εργασία τους σπουδαστές αυτούς. Και θα πρέπει να έχουμε και τους ελέγχους υπό το άρθρο 31 για την ε, συλλογή και παρακολούθηση των ε, προσωπικών αυτών δεδομένων. Είναι επίσης πολύ σημαντικό μέσω της ε, συνολικής προσέγγισης να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλους τους τομείς ε, και, για τους, ε, και επί τη βάση αναπηρίας και επί τη βάση φύλων. Δηλαδή με οριζόντιο τρόπο αν θέλετε. Φυσικά το ίδιο ισχύει για την αγορά εργασίας. Πρέπει να έχουμε επαρκείς ε, διατάξεις και ευέλικτες διατάξεις, επί παραδείγματι στην φάση της επιλογής, ώστε να μπορεί κανείς μέσω της εργασίας, μάλλον η εργασία του να το επιτρέπει να φροντίζει και τα παιδιά του. Θα πρέπει λοιπόν και οι γυναίκες να έχουν κάθε δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους προκειμένου να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν να υποστηρίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι γυναίκες αυτές. Ας δούμε αν έχουμε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Βανχέης. Αναδείξατε πολλά σημαντικά θέματα, ιδιαίτερα στον τομέα της αγοράς εργασίας. Χρειαζόμαστε διατονομιακή ε, νομοθεσία και συνεργασία όλων, κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Σας ευχαριστώ πάντως που αναδείξατε το ζήτημα. Τελευταία μας ε, ομιλήτρια, κυρία Πρόμπστ. Γιούλια, έχετε το λόγο. Gut, erstmal guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. γνώμη υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ένα μπουκάλι με νερό εμποδίζει την διερμηνέα. Ε, ακούω λοιπόν εδώ καιρό τους συναδέλφους μου και έχω την αίσθηση ότι σχεδόν ανταγωνίζονται οι χώρες για το ποια κάνει τις περισσότερες διακρίσεις. Ε, ομολογώ ότι μου προκάλεσε έκπληξη. Είμαι κοφή, οπότε για μένα η νοηματική γλώσσα δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που έμαθα όταν ήμουν 17 χρονών. 90% των παιδιών με προβλήματα ακοής μεγαλώνουν σε οικογένειες με γονείς που ακούν κανονικά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο λοιπόν για αυτούς να έχουν πρόσβαση σε μια εναλλακτική γλώσσα, εννοηματική γλώσσα πολύ συχνά δεν προσφέρεται, δεν τους προσφέρεται, που σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά και οι νέοι άνθρωποι σε πολλές, φορές, σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν. Ό,τι είπατε για τα άτομα με, ε, διανοητική, με διανοητικά προβλήματα σε σχέση με την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά συνδέεται με γυναίκες με προβλήματα ακόης. 52% των γυναικών που έχουν προβλήματα ακοής στην Γερμανία, σύμφωνα με μία έρευνα, έχουν πέσει θύματα α, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Απλούστατα γιατί δεν μπορούν να πούν τι του συνέβη, γιατί δεν έχουν μια γλώσσα να επικοινωνήσουν αυτό το οποίο του συνέβη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει μια hotline, μια γραμμή, τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για γυναίκες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι γυναίκες με προβλήματα ακοής έχουν μόνο ένα παράθυρο από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με κάποιο άτομο που να τους καταλαβαίνει, ενώ οι υπόλοιπες γυναίκες έχουν 24 ώρες την ημέρα στην διάθεσή τους και για να μπορέσει μια γυναίκα με προβλήματα ακοή να χρησιμοποιήσει αυτήν την συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή πρέπει να φορτώσει ένα λογισμικό πρόγραμμα που θα τη επιτρέψει να έχει πρόσβαση. Με άλλα λόγια, αν δεν έχει πρόσβαση στην κατάλληλη τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την hotline καθόλου. Πρέπει να έχεις αυτό το software στον υπολογιστή σου, πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως σε μια δύσκολη περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την τεχνολογία που είναι απαραίτητη. Όταν οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας στο σπίτι τους, προβλήματα οικογενειακής βίας και θέλουν να πάνε σε κάποιο από τα καταφύγια, είναι δύσκολο να βρουν έναν διερμηνέα νοηματική. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικό οι γυναίκες αυτές να μπορούν να επικοινωνήσουν, να, να πούν τι τους συνέβη όταν φτάνουν σε αυτά τα καταφύγια. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα αφορά τις γυναίκες με αναπηρία. Αν πρέπει να πάνε σε μια κρόαση, για παράδειγμα, συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε διερμηνείς νοηματικής και μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για αυτές να εξηγήσουν ποια ήταν η εμπειρία τους και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάστασή τους χωρίς την μεσολάβηση ενός διερμηνέα νοηματικής. Θέλω απλώς να σηκωθώ για να δείτε ότι είμαι έγκυος. Αυτό είναι το πρώτο μου παιδί, είναι η πρώτη μου εγκυμοσύνη. Ήταν δύσκολη η διαδικασία. Μπορώ κατά κάποιο τρόπο να, μιλήσω, αλλά πολλές γυναίκες με προβλήματα ακοής δεν μπορούν καθόλου. Αν λοιπόν η επικοινωνία μια γυναίκα με προβλήματα κόη περιορίζεται μόνο στον διερμηνέα τη νοηματικής, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολα στην επικοινωνία τη με τον γιατρό ή το νοσηλευτικό προσωπικό. Και είναι καθαρά στην ευθύνη των γυναικών αυτών με προβλήματα ακοή να βρουν έναν διερμηνέα αν προκύψει κάτι επίγον και πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Πολύ συχνά μπορεί να μην μπορώ να έχω έναν διερμηνέα νοηματική την τελευταία στιγμή. σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή όπου μπορείς σε, επίγο σε επίγοντα περιστατικά, σε επίγουσες περιπτώσεις να βρεις έναν διερμηνέα νοηματικής, αυτό όμως δεν ισχύει παντού στη Γερμανία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος νόμος που να ορίζει πώς ε, πληρώνονται οι διερμηνεί αυτοί. Και με την ασφάλεια μου κάθε φορά υπάρχει συζήτηση, υπάρχει καυγάς για το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Υπάρχει ένα νομικό κενό, με άλλα λόγια. Αν εγώ ως άτομο με προβλήματα ακοής πάω στο γιατρό αλλά οι γονείς μου μπορούν να ακούν και πρέπει να επικοινωνήσω με τον γιατρό φυσικά, τότε εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μιλήσω για τον αυτό μου, είναι οι γονεί μου που θα πρέπει να επικοινωνήσουν για μένα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική. Περίπου 80.000 άτομα με προβλήματα κοής στην Γερμανία. Μόλις 3% έχουν το απολυτήριό τους. Δεν υπάρχουν στοιχεία σε ό,τι αφορά το ποσοστό των γυναικών μέσα σε αυτό το 3% που σας ανέφερα. αν, ε, αν κάποιος θέλει να συνεχίσει τις σπουδέ του, τα έξοδα διερμηνίας νοηματικής δεν καλύπτονται. Πράγμα που σημαίνει ότι αν αποφασίσει να συνεχίσει σπουδέ σου πρέπει να το κάνεις χωρίς διερμηνία νοηματικής. Ένα άλλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση είναι οι καθηγητές με προβλήματα ακοής. Με συγχωρείτε, αυτό που ήθελα να πω είναι οι καθηγητές για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Όταν ένας φοιτητής, για παράδειγμα, θέλει να συνεχίσει τις σπουδέ του, δεν υπάρχει προϋπόθεση διερμηνίας νόηματική σε κάποια πανεπιστήμια. Προσφέρεται, σε καμία περίπτωση δεν είναι ο κανόνας όμως αυτός. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει δυνατότητα να εκπαιδευτούν οι καθηγητές για να διδάσκουν άτομα με προβλήματα ακοής. Είναι λίγο δύσκολο για μένα να συγκεντρωθώ γιατί το μωρό μου κλωτσάει καθώς σας μιλάω. Επιστρέφοντας λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα για τα επίγοντα περιστατικά στη Γερμανία, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμός που μπορείς να καλέσεις. Και πάλι όμως υπάρχει, έχει τη δυνατότητα μέσω του υπολογιστή σου, αν έχει ένα συγκεκριμένο λογισμικό, αν έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε σε περίπτωση μιας επίγουσα περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε πρέπει να έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε κάποιον να μπορεί να μας βοηθήσει. Όλες οι επιλογές μας είναι μέσω του διαδικτύου. Και αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι γιατί η Γερμανία δεν μπορεί να έχει ένα σύστημα ας πούμε, μέσω μηνυμάτων στο κινητό. Αν για παράδειγμα το σπίτι μου πάρει φωτιά, δεν μπορεί να με απασχολεί πώς θα συνδεθώ στο διαδίκτυο. Δεν είναι φυσιολογικό. Ή αν βλέπω μια ταινία στην τηλεόραση, ή αν παρακολουθώ τις εκλογές, υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσω διερμηνία στην νοηματική, αλλά και πάλι είναι μέσω του διαδικτύου. Όλες οι επιλογές για τα άτομα με προβλήματα ακοή είναι μέσω του διαδικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα που είναι μια μεγαλύτερη ηλικία και έχουν προβλήματα ακοή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία, δεν γνωρίζουν πώ να τη χρησιμοποιήσουν. για πολλούς ανθρώπους είναι και πρακτικό το ζήτημα. Η οθόνη είναι πάρα πολύ μικρή, απλούστατα δεν μπορούν να βλέπουν τον διερμηνέα νοηματικής. Έχω την αίσθηση ότι γυναίκες με προβλήματα κοής, ιδίω στην Γερμανία, δεν έχουν και πολύ μεγάλη πρόσβαση σε αυτού του τύπου την τεχνογνωσία. Χρειάζονται βοήθεια κάποιον να τους εξηγήσει, κάποιον να τους εκπαιδεύσει. αυτό που μας ενώνει όλους επί της ουσίας είναι ένα ζήτημα εκπαίδευσης και ένα ζήτημα επικοινωνίας. Θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότερες διακρίσεις εναντίον των γυναικών με προβλήματα κοής σε σχέση με τους άντρες με προβλήματα κοής. Αυτό που επίσης χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες με προβλήματα ακόης και τις ανάγκες τους. Πρέπει να έχουμε περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διάθεσή μας, περισσότερη βοήθεια. Και αν θέλω εγώ να χρησιμοποιήσω κάποια από αυτές τις υπηρεσίες δεν μπορεί να πρέπει να περιμένω τρει ή τέσσερι εβδομάδες για να βρεθεί διερμηνέας νοηματικής. Υπάρχουν τόσα πολλά οργανωτικά προβλήματα και τεχνικά ζητήματα που τελικά δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Προσπάθησα απλά να θίξω τα πιο σημαντικά ζητήματα και ολοκληρώνω την ομιλία μου εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Γιούλια λέει η Πρόεδρος. Μίλησες πολύ για θέματα επικοινωνίας ε, και ευαισθητοποίησης και ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι κάτι κάναμε επ' αυτού σήμερα. Θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια προτού συνεχίσουμε με το διάλογο να μας ε, δώσει μια σύντομη εικόνα παρακαλώ. Η κυρία Φεραγούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να καλασορίσω όλους τους καλεσμένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπαν και όλα αυτά τα στοιχεία θα τα λάβουμε υπόψη μας στην γνωμοδότηση. Ε, εγώ στην Επιτροπή Γυναικών Είχα ήδη συζητήσει από την προηγούμενη εντολή το θέμα μιας τέτοιας ε, γνωμοδότησης. Ε, δουλέψαμε πολύ με την Αναπελάιθ και όλους τους οργανισμούς και ενώσεις ε, στην Ευρώπη. Και εδώ προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να φέρουμε το θέμα στην επιφάνεια. Των γυναικών δηλαδή με αναπηρία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το να είναι εμφανές το θέμα αυτό. Κατά δεύτερον, να υπάρχουν κοινοί δείκτες στα κρατημέλη. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική επί του θέματος λαμβάνει υπόψη της και το θέμα των φύλων, αλλά πρέπει να έχουμε κοινούς δείκτες. Διότι έχουμε δυσκολίες σε κάποια κράτη-μέλη γιατί δεν αποφασίζουν όλα τα κράτη κατά τον ίδιο τρόπο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων επί τη βάση των αναπηριών ή του φύλου. Χρειαζόμαστε λοιπόν δουλειά σε όλους τους τομείς, στο ε, θέματα εργασίας. Έχουμε τη σύμβαση, είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πόσο μάλλον αν έχουν και αναπηρίες και πρέπει αυτό το θέμα να το καλύπτουμε διότι η εργασία δεν είναι απλώς μια πηγή εσόδων. Είναι ένα μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης, ένταξης. Επομένως είναι θεμελιώδους σημασίας. Προφανώς τα θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτισης. Στα θέματα παιδείας δεν δουλεύουν όλα τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής παιδείας, που είναι θεμελιώδες ώστε να έχουμε μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων και που να πιστεύουμε πραγματικά στην ενεργό και ίση συμμετοχή όλων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα που δουλεύουν στα θέματα συμμετοχικότητας, τα λίγα αυτά κράτη-μέλη, και όχι σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με αυτό, σημειώνουμε ότι οι γυναίκες με αναπηρία και γενικώ οι άνθρωποι με αναπηρία αφήνονται χωρίς πλήρη προσβασιμότητα από τα συστήματα παιδεία στην άκρη, στο περιθώριο. Χρειάζεται λοιπόν η πρόσβαση για να μπορεί κανείς να συνεχίσει να παρακολουθεί τα προγράμματα αυτά. Επομένως και στον τομέα της παιδείας υπάρχουν θέματα ίσων δικαιωμάτων. Στα θέματα υγείας ελέγχθη μας λείπουν οι ειδικεύσει, οι ειδικότητε των ε, επαγγελματιών που θα βοηθούν και θα υποστηρίζουν τους ανθρώπους και τις γυναίκες με αναπηρία. Χρειάζεται συγκεκριμένη κατάρτιση, χρειάζεται πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, χρειάζεται ενημέρωση για τις γυναίκες, χρειάζεται σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παιδεία για να μπορεί να είναι σε θέση να αποφασίζει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να προστατεύουμε την ε, οικογενειακή ζωή Συμφωνώ απολύτως ότι η στήρωση και οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ε, αναπαραγωγικής ικανότητας ε, είναι παραβίαση θεμελίως δικαιώματος. Χρειάζεται να εξασφαλίζεται το δικαίωμα πλήρους σεξουαλικής ζωής και βεβαίως μητρότητας. Χρειάζεται λοιπόν μια αλλαγή σχεδιασμού και εμβάθυνση σε όλα τα θέματα αυτά. Ε, τα, τα θέματα πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Χωρίς τέτοια πρόσβαση σήμερα έχουμε απόλυτη διακρίση. Είναι προφανές. Χρειάζεται λοιπόν προσαρμογές για τη γλώσσα των ανθρώπων με προβλήματα ακοής, ε, για τις τεχνολογίες που μας χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση και οι άνθρωποι αυτοί. Και υπάρχει και θέμα δημοκρατικής Συμμετοχή έλλειμμα αν θέλετε δημοκρατικότητας υπό την έννοια αυτή. επομενω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το, την ίση πρόσβαση στο δικαίωμα ψήφου γιατί χωρίς αυτό η δημοκρατική συμμετοχή δεν έχει νόημα και η δημοκρατική συμμετοχή, η ίση συμμετοχή είναι και αυτό εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι για τις γυναίκες με αναπηρία στην περίπτωση μητρότητα θα έπρεπε να έχουμε διευρυμένη άδεια μητρότητας. Τώρα, είναι, δεν υπάρχει αφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα αυτά. Το να μην τα φροντίσουμε αυτά τα θέματα σημαίνει μεγαλύτερη απομόνωση σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα μειονεκτήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία και γι' αυτό μας χρειάζονται εξτρατείες ευαισθητοποίηση στα κράτη-μέλη. Από τις οποίες εξτρατείες διαφωτίζεται, εμπλουτίζεται αν θέλετε το σύνολο της κοινωνίας. Και δυστυχώς ένα άτομο με αναπηρία έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι θύμα κρούσματος βίας και βίας επί τη βάση του φίλου. Χρειάζεται λοιπόν να εντάσσεται η, ένταξη, η διάσταση του φίλου και των αναπηριών σε όλες τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα θέμα που εγκρίναμε πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες, δεν θυμάμαι καλά, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα, που ήταν μια ευκαιρία. Ήταν μια ευκαιρία, διότι το Κοινοβούλιο είχε δεσμευτεί στην κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή έκανε μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, λογική. Εγώ ήθελα περισσότερα. Ε, όμως το κοινοβούλιο ήταν διαρρεμένο. Δώσαμε μεγάλη μάχη μεταξύ μας. Ε, ελπίζει κανείς και θα ελπίζει κανείς ότι στον τριμερή διάλογο μπορούμε να βελτιώνουμε πάντοτε τα θέματα αυτά, οποιαδήποτε πρόταση. Ε, και γι' αυτό κάθε τέτοια προσπάθεια είναι απολύτως απαραίτητη και μας βοηθάει στα θέματα δικαίου, στα θέματα ίσης ε, ευκαιρίας, ε, συμμετοχικότητας, να προχωρούμε λίγο ακόμα προς τα εμπρός. Σας ευχαριστούμε. Την περιμένουμε με ανυποπονησία την εκθέσή σας, γιατί θα είναι πολύ σημαντική και θα είναι σημαντικό επειδή έχουμε να από την Επιτροπή μας. Έχω ε, τρεις ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο τρία μέλη της Επιτροπής. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 10.30. Ε, Κύριε Μόβάη, μια τεχνικής φύσους ε, ερώτηση. Υπάρχει διερμηνία από τα Ουγγρικά. Η Πρόεδρος δυστυχώς όχι. Σήμερα δεν είχε προβλεφθεί η διερμηνία από τα ογκρικά. Η ομιλήτρια μου φαίνεται προβληματικό το ότι σε μια συνεδρίαση όπου συζητούμε την ισότιμη μεταχείριση της ευκαιρίας δεν έχουμε την διερμηνία για τη γλώσσα μου. Η Πρόεδρο, το συγγνώμη, με ενημέρωσε η υπηρεσία διαρμηνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι για να καλυφθεί η διαρμηνία για τους άλλους ομιλητές, τους προσκεκλισμένου μας, δεν υπήρχε δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα οκλικά, πάντως ζητώ συγγνώμη. <coughs> η ομιλητρία. Κυρία Μορβάη, τέλος πάντων να συζητήσουμε το θέμα το πιο σημαντικό που συζητούμε σήμερα. Ήταν πολύ χρήσιμο κατά την άποψή μου ότι ακούσαμε την εμπειρία ατόμων, γυναικών με αναπηρία, τις προσωπικές τους δηλαδή εμπειρίες ανθρώπων που πλήττονται από αυτά τα προβλήματα. Ε, θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμο να ακούσουμε τέτοιου τύπου μαρτυρίες. Ιδιαίτερως θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσκεκλημένη μας που μας μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οικοφή. ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβασή τους στι υπηρεσίες υγείας, το τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση μια ε, επίγοντο ιατρικού προβλήματος, καθώς επίσης και τα προβλήματά τους στην πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης. Υπάρχει πρόβλεψη για διερμηνία νοηματικής στους φοιτητές που τη χρειάζονται. Υπάρχει καν αυτή η πρόβλεψη, πρόβλεψη, υπάρχει ε, τέτοια πρόβλεψη για τα νοσοκομεία. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω για άλλες μορφές ε, αναπηρίας ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που ε, οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα οι τυφλοί. Αυτό που δεν κατάλαβα και πολλοί από τις παρουσιάσεις είναι τι εννοούμε ακριβώς όταν μιλούμε για την παραβίαση του δικαιώματος στην ψήφο. Αναφέρθηκε ότι κάποια εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν έχουν, το δικαίωμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ψήφο. Μιλούμε για τα άτομα με διανοητική αναπηρία εδώ, μιλούμε για κάποιο άλλο είδους πρόβλημα, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουν το δικαίωμα στην ψήφο. Ε, ένα θεμελιώδες. Ε, ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πραγματικά θα ήθελα να μου το εξηγήσετε περισσότερο, να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να ακούσουμε τις, ε, την εμπειρία που έχουν οι γυναίκες οι οποίες φροντίζουν κάποιο παιδί με αναπηρία στο σπίτι τους. συζητούμε πολλά διαφορετικά ζητήματα που συνδέονται με τη μητρότητα. Το ένα ζήτημα είναι η μητρότητα των ιδίων των γυναικών με αναπηρία. Το άλλο ζήτημα είναι πώς υποστηρίζουμε τη μητρότητα κάποιες γυναίκας, που το παιδί της έχει αναπηρία. Και σε αυτό το θέμα θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η προσέγγιση των κρατών μελών. Η πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά έχουμε έξι λεπτά στη διάθεσή μα και έχω ακόμα δύο ομιλητέ. Η ομιλήτρια, κλείνω. Το επόμενο ερώτημα είναι ποιοι οικονομική πόροι είναι στη διάθεση των γυναικών αυτών ε, στα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Τχάντ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλε τις εισηγήτριες για τις ενδιαφέρουσες ε, τοποθετήσει τους ε, να σας συγχαρώ και την κυρία Πρόπστη για την μητρότητά της θα έχετε, είμαι σίγουρη, μια υπέροχη εμπειρία. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό αρκετές φορές. Των γυναικών που αντιμετωπίζουν αναπηρίες και το, ε, το πόσο πάρα πολύ συχνά είναι θύματα διακρίσεων γιατί οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν μάλλον οι γυναίκες ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξ αρχής ε, για την απορρόφωτησή τους ε, ή στην αγορά εργασίας, πόσο μάλλον οι γυναίκες με αναπηρία. Δυστυχώς όταν έχουμε ένα νομοθέτημα σημαντικό που αφορά στις, ε, στα ίσα δικαιώματα στους ανθρώπους με αναπηρία όπως κάναμε πριν από κάποιες εβδομάδες ε, για την ε, οδηγία για την προσβασιμότητα που αναφέρθηκε νωρίτερα εδώ όπου η Επιτροπή είχε υποβάλει μια θαυμάσια πρόταση και το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να προχωρήσει το πράγμα προς τα εμπρός, δεν κατάφερε να συμφωνήσει στάθηκε, ε, φάνηκε να είναι κατά της ε, ε, οδού, της πρόοδου που θα μας οδηγούσε μια βελτίωση της κατάστασης για τους ανθρώπους με αναπαρία. Χρειαζόμαστε ίσες συνθήκες, ισότιμες συνθήκες για όλους και γι' αυτό είχαμε υποβάλει και μια γνωμοδότηση της οποίας ήμουν εισηγήτρια για την για τις γυναίκες με αναπηρία στον, στην οικονομία, στον οικονομικό τομέα. Το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην απορρόφηση από την, από την αγορά εργασίας. Είναι πολύ δύσκολο να αναφέρει κανείς όλα τα σημαντικά θέματα βέβαια. Κάτι που μου έρχεται στο νου πάντως έχοντας ακούσει όλα αυτά είναι το θέμα των στατιστικών δεδομένων χρειαζόμαστε για την ίδια δουλειά να έχουμε τον ίδιο μισθό. Χρειαζόμαστε μια χαρτογράφηση, μια απεικόνηση της διαφοράς που έχουμε σήμερα. Πόσο μάλλον για τις ε, γυναίκες μια αναπηρία. Και μου έρχεται στο νου το Ινστιτούτο Ισότητας που έχουμε, λέει, ομιλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αν μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση. Εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι επιτάπητος. Και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή την ώρα που νομοθετούμε και στο Κοινοβούλιο για να συμπεριλάβουμε, να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ κυρία Ράνκε το συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα για όλη τη διάρκεια τη ακρόαση. Είχα ε, μια επανειλημμένη υποχρέωση σε άλλη επιτροπή. Τρία θέματα θέλω να θέξω που σχετίζονται με την έκθεση. Πρώτα απ' όλα η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ ε, που ήδη αναφέρθηκε πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί στην πράξη και για να γίνει αυτό πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Έχουμε διαπιστώσει ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο δεν προχωρά και χρειάζεται να ασκήσουμε την πίεσή μας έτσι ώστε τελικά να οδηγηθούμε σε ε, ουσιαστική εφαρμογή της συνθήκης αυτής και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Δεύτερον, το ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι, έχουμε αρμοδιότητα νομοθε... νομοθέτησης σε ζητήματα όπως αυτά που σχετίζονται με την αγορά της εργασίας, ε, με την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ε, επομένως, οφείλουμε να εκφράσουμε την άποψή μας με μεγαλύτερη ένταση γιατί ε, είναι, ε, εμείς προωθούμε κάτι το οποίο είναι το σωστό. Ε, και το τρίτο. Είναι ένα άλλο εργαλείο που έχουμε στη διαθεσή μα είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η χρηματοδότηση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μπορούσε να προωθήσει τα ζητήματα αυτά. όχι μόνο η χρηματοδότηση για ζητήματα ισότητα, αλλά επίση και τα διαρθρωτικά ταμεία, στα, στα, στα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για έργα που θα καταστήσουν τις υποδομές περισσότερο προσβάσιμες ή ισότιμα προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ε, πιέσουμε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αυτό που μας λένε ότι βεβαίως ε, εμείς είμαστε όλοι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά δεν έχουμε πόρους στη διάθεσή μας. με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι μπορούμε να πιέσουμε για την πρακτική εφαρμογή αυτών των ε, ε, θεμάτων, αυτών των ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Η Πρόεδρος, ε, ορισμένοι από τους διερμηνείς είναι, βρίσκονται σε άλλες συνεδριάσεις αμέσως μετά. Επομένως, δυστυχώς, και 10.30 πρέπει να διακόψουμε την παροχή υπηρεσία της διερμηνίας. Ε, θα προτείνω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μονάχα στα αγγλικά, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές, τον ένα μετά τον άλλο, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Καλό, καλή ημέρα από εμάς. Um, especially giving us the possibility to, to talk uh, a little more. Um, can, I, can I just make one um, additional comment? Just 4% of all disabled people are